Γκρίνω τα πρακτικά. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια μας διάταξη είναι η δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την οικονομική κρίση. Συνάδελφοι, τουλάχιστον θα έχω την χαρά μου, τη χαρά να μιλήσω στην άδεια αίθουσα. Είστε πολύ πεπειραμένοι από αυτή την άποψη. I have spoken to both presidents, Van Rompuy and Barroso. Καλωσορίζω τους δύο. Ε, μάλλον ε, θέλω να μιλήσω με τους δύο προέδρους ε, Van Rompuy και Μπαρόζο και θα τους ενημερώσω για τα αποτελέσματα της σημερινής μας συζήτησης στην Ολομέλεια. Την στην αναρτήρια ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ομιλία μου, συγγνώμη, στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, υποστήριξα ότι ένα ολοκληρωμένο και αποφασιστικό πακέτο θα πρέπει να είναι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων ε, για να ξεπεραστεί η ευρωπαϊκή κρίση και ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να συνεργαστούν. Θυμήσατε στο Συμβούλιο ότι είμαστε το Ευρωκοινοβούλιο της Ευρωζώνης και γι' αυτό και καλωσορίζω ότι ανάμεσα στην ε, Κυριακάτικη Διάσκεψη Κορυφής και την Αυριανή θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να συζητήσουμε τις μέσο και μακροπρόθεσμες λύσεις που είναι επιτάπητος. Το συμπέρασμά μου είναι ότι υπάρχουν τρία επίγοντα θέματα το, η μείωση του χρέους της Ελλάδας, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς και με, σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να α, γίνει εθελοντική αναδιάρθρωση ή ανακεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών όπου ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις στο ΕΚΟΦΗΝ των 27 χωρών μελών όπως οι απαιτήσει κεφαλαίου και η καταλληλότητα που θα ανέβει στο 9%, το πώς ε, θα συγκεντρωθούν χρήματα από τι αγορές μέσω των εθνικών προπολογισμών και του EFSF. Αυτά θα πρέπει ακόμα να αποφασιστούν και πιστεύω πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει λόγο επ' αυτών. Και το τρίτο σημείο είναι η δημιουργία ενός προστατευτικού τείχους γύρω από τις οικονομίες που ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το Συμβούλιο αύριο θα αποφασίσει για την ενίσχυση του EFSF επιτρέποντάς του να μπορεί να συνεργαστεί με μηχανισμούς ασφάλειας. Υπάρχουν ακόμα δύο εκκρεμή θέματα όσον αφορά το προστατευτικό τείχος, η δημιουργία δηλαδή ενός χήματος ειδικού στόχου και η δημιουργία ενός ταμείου με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μεσοπρόθεσμα χρειάζεται να δοθεί χρόνος για την ενίσχυση του, μάλλον για το ενισχυμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ή διαφορετικά το πακέτο των έξι οδηγιών, που είναι όλα κίνητρα για την ανάπτυξη. Ε, ορισμένες αρμοδιότητες ίσως να είναι εθνικού χαρακτήρα, αλλά τα περισσότερα κρατημέλη συμφωνούν ότι πρέπει να συντονιστούμε πολύ καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σημαντικό ερώτημα είναι πώς θα κινήσουμε όλα αυτά τα θέματα από το διακυβερνητικό πλαίσιο στο κοινοτικό. Είναι σημαντικό οι βράχοι και οι μέσο πρόθεσμες λύσεις να ανατεθούν στα ευρωπαϊκά όργανα. Πιο μακροπρόθεσμα γίνονται συζητήσεις για μια πιθανή αλλαγή στη συνθήκη. Το ερώτημα είναι τι είδους αλλαγή αναμένουμε. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιασδήποτε αλλαγές. Μακροπρόθεσμα χρειάζεται να καταλήξουμε σε συμπεράσματα από αυτήν την κρίση και να προβληματιστούμε για το μέλλον της Ένωσης. Σίγουρα θέλουμε να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους παγκόσμιους παίκτες. Και η κρίση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να ενεργήσουμε γρήγορα. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια κατάσταση ενότητας που στην ουσία όμως είναι ένας, ένα είδος κατακαιρματισμού. Το ξέρουμε αυτό στη θεωρία, αλλά στην πράξη μιλάμε για την Ένωση, αλλά ε, βασικά τις πολιτικές μας σχηματίζουμε σε εθνικό επίπεδο. Η Ένωση μοιάζει να είναι ένα όνειρο, ενώ το κράτος έθνος είναι αυτό το οποίο λειτουργεί και αποφασίζει. Αυτή είναι η αδυναμία μας και χρησιμοποιείται κατά των κοινών μας στρατηγικών ευρώντων. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ισχυρή σε έναν σύγχρονο και πολύπλευρο κόσμο. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο η κοινή αγορά αλλά είναι μια συνεπής και συνεκτική πολιτική ιδέα, εικόνα που μπορεί όχι μόνο να ξεπεράσει κρίσεις, αλλά να έχει και αντίκτυπο στον σύγχρονο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, okay. Now we go to the... Οπότε τώρα περνάμε στις δηλώσεις των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κόριν Βόρτμαν Κόλ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα εδώ πέρα στο Στρασβούργο ο κύριος Φαν και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, βρίσκονται στις Βρυξέλλες για να λάβουν αύριο τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για να βγει η Ευρώπη από την κρίση. Έχει λοιπόν κηρυχθεί απόλυτη σιωπή ασυρμάτου και αναμένουμε τις αποφάσεις. Οπότε, σε τι βασιζόμαστε, σε άρθρα στον τύπο, σε κάποια έγγραφα της συνεδρίασης, αλλά επίσης κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πάρα πολλέ ανησυχίε και πάρα πολλή αβεβαιότητα στους πολίτες μας, γιατί από ό,τι φαίνεται η κρίση μόνο επιδεινώνεται και οι οικονομικές προοπτικές επιδεινώνονται. Ανησυχούν οι πολίτες μας για τις δουλειέ τους, για τις συντάξει τους και γι' αυτό θα ήθελα εξ ονόματο της ομάδας μου να καλέσω τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων να έχουν θάρρος, να μην κάνουν μεσοβέζικες λύσεις, αλλά μια συνολική αντιμετώπιση της κατάστασης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις χρηματαγορές και να υπερασπίσουμε το ευρώ από την ε, επίθεση την οποία δέχεται. Είχαμε μέχρι στιγμής πάρα πολλές μεσοβέζικες λύσεις και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αποδείξουμε πως η Ευρώπη είναι σε θέση να κάνει αυτά που πρέπει. Είναι πλέον 12 και 5. Κύριε Πρόεδρε, η αιτία της κρίσης βρίσκεται στα κράτη-μέλη, αλλά τα προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη μας αγγίζουν όλους. Έχουμε ένα κοινό νόμισμα, από το οποίο υποφελούμαστε όλοι, κάθε χρόνο. Και αυτό μας υποχρεώνει να είμαστε αλληλέγγυοι και να αναζητήσουμε λύσεις. Η ενίσχυση του EFSF και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο κεφαλαιοποίησης των τραπεζών είναι απολύτως απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα με μία μόνιμη λύση και να ε, αποκατασταθεί η ηρεμία στις χρηματαγορές. Το EFSF πρέπει επιτέλους να αποκτήσει τη δύναμη πυρός ενός μπαζούκα και πολύ περισσότερα κονδύλια. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά εάν μπλοφάρουν οι αγορές για το ευρώ πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε αυτή την πλόφα για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά μας. Κύριε Πρόεδρε, η ασφάλεια, η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ώστε χώρες και τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας γιατί ο κίνδυνος εδώ πέρα μετάδοσης της κρίσης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πρέπει να φροντίσουμε να μην καταρρεύσουν και οι τράπεζες γιατί ένα σταθερό οικονομικό σύστημα έχει σημασία για την οικονομική ζωή και σταθερότητα και για τις δουλειές μας. Βεβαίως, οι τράπεζες κατά κύριο λόγο είναι οι ίδιες υπεύθυνες για να προσελκύσουν κεφάλαια. Το Ταμείο αυτό θα είναι μόνο η λύση ανάγκης και επίσης δεν θα τις ε, δίνει και κίνητρα για την ανεύθυνη συμπεριφορά τους, αντιθέτως θα πρέπει να συνοδευτεί από μία δέσμευση για αναδιάρθρωση της ε, λειτουργίας τους. Αλλά είναι απαράδεκτο, το αντιλαμβάνεστε, για τους φορολογούμενους να δίνουμε τα λεφτά τους για να θειασώσουμε τις ε, τράπεζες. Οπότε θα πρέπει να τεθούν κανόνες χρηματαγορές. Επίσης, το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ένας ισορροπημένος φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών για να μπορέσει να λειτουργήσει και ένας φόρος επί των τραπεζών για να αντιμετωπιστεί ακριβώς η κρίση. Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζουμε τις αποφάσεις της ε, Κυριακής μας πέρασε για να επιταχυνθούν οι έξι οδηγίες και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για να βάλουμε τα του οίκου μας σε τάξη. Και πρέπει να προχωρήσουμε παραπέρα, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη και άρα είναι σημαντικό αύριο να γίνουν σημαντικά βήματα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωζώνης. Πρέπει επίσης να περάσει το σύμφωνο Ευρώ-ΣΥΝ και οι προτάσεις της ε, Κομισιόν λένε πως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση στον προπολογισμό των κρατών μελών. Και αυτό χρειάζεται. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση στο ευρώ και στην εσωτερική μας αγορά και αλλαγή της συνθήκης θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος. Αλλά σημαντικό είναι να γίνει αυτή η συζήτηση με τους πολίτες μας γιατί έχει κρίσιμη σημασία να στηρίζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα οι πολίτες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, ο κύριος Μάρτιν Σούλτς για τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είδαμε την έκθεση, κύριε Πρόεδρε, και θα ήθελα να πω πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ετάρτης ίσως πραγματικά αξίζει το επίθετο ιστορικό. Δεν χρησιμοποιώ συχνά αυτή τη λέξη, αλλά πιθανώς αυτό το οποίο θα συμβεί αύριο στις Βρυξέλλες έχει ιστορική σημασία. Γιατί το ερώτημα πού πηγαίνει η Ευρώπη μάλλον θα κριθεί αύριο. Έχω ασκήσει πάρα πολύ συχνά κριτική το ότι έχει τρία μέρη η Ευρώπη. Ένα γαλλογερμανικό διευθυντήριο, την υπόλοιπη Ευρωζώνη και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδιαίτερη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ο κατακριματισμός της Ευρώπης σε διαφορετικές δομές είναι ήδη από μόνο του ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους. Καταστρέφει την κοινωτική μέθοδο και στο τέλος δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία η εξάρτηση όσων δρούν εντός της Ευρωζώνης από την εσωτερική κατάσταση της χώρας τους είναι τόσο δραματική ώστε ο καθένας ο οποίος κάθεται γύρω από αυτό το τραπέζι σκέφτεται μόνο την εθνική του κατάσταση αντί να επιδείξει κοινοτικό πνεύμα και να αποτελέσει βάση της ε, δράσης του το κοινό συμφέρον. Το είδαμε στη Σλοβακία, το είδαμε στη Γερμανία, το βλέπουμε σε κάθε χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και μην ξεχνάμε ότι στο Συμβούλιο των 17 του Ευρώ υπάρχει ομοφωνία και απαιτείται ομοφωνία και ε, αποτελούμε μία από τις ισχυρότερες νομισματικές ζώνες του κόσμου ανεξαρτήτως των παιγνίων των μικροπολιτικών. Οπότε θα πρέπει να έχουμε τα κοινά μας εκείνα θεσμικά όργανα τα οποία θα μπορούν να επιβάλλουν την κοινή μας πολιτική. Δεν χρειάζεται όμως να εφεύρουμε τίποτα το καινούριο. Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα δύσκολο δρόμο γιατί εδώ πέρα διακινδυνεύει η εμπιστοσύνη των αγορών στην βιωσιμότητα των επενδύσεών τους στην Ευρώπη και η εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εάν μπορούν να τα διαχειριστούν αυτά αποτελεσματικά. Αυτή η εμπιστοσύνη διακυβεύεται εδώ και 1,5 χρόνο ο κανόνας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι διακηρύσουμε και δεν εφαρμόζουμε. Το παίρνουμε πίσω, το ξαναγυρνάμε από εδώ από εκεί, το ξανανακοινώνουμε και πάλι δεν εφαρμόζουμε τίποτα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είδαμε πως συναντήθηκε ο κύριος Σαρκοζή με την κυρία Μέρκελ και τι είπανε, είπανε πως πάλι τα ίδια, συμφωνήσαμε. Και όμως Κυριακή βγαίνουν ε, από το Συμβούλιο Μέρκελ και και δίνουν συνέντευξη τύπου. Για τι πράγμα, για τα πράγματα στα οποία δεν συμφώνησαν. Είναι όμως σαφές στον καθένα ποιο είναι το διακύβημα εδώ πέρα και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Είναι το ύψος του κουρέματος. Και το ύψος αυτού του ψαλιδίσματος εξαρτάται από το πόσο πολύ πλήττονται οι γαλλικές τράπεζες από αυτό. Αυτές πλήττονται περισσότερο και γι' αυτό το γαλλικό κράτος ξέρει πως εάν γίνει αυτό θα πρέπει να σταθεροποιήσει τις τράπεζές του, το αναφέρατε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει από τον εθνικό του προϋπολογισμό το γαλλικό κράτος, γιατί απειλεί η κυρία Ρέντινγκ. Οπότε θα προσφύγει στο EFSF. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πέρα δύο μοντέλα το γαλλικό και το γερμανικό. Και πάνω σε αυτό δεν συμφωνούν. Αντί λοιπόν να έχουμε αυτό το παζάρι θα έπρεπε να μπουν σε μία αίθουσα και να μην βγουν μέχρι να βγει από την καμινάδα λευκός καπνός. Θα πρέπει για πρώτη φορά να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να πω κάποια πράγματα για πιθανή αλλαγή της συνθήκης. Διαβάζω, ακούω πώς πρέπει να αλλάξει η συνθήκη, πώς έχει ξεκινήσει ήδη μια ομάδα εργασίας με τον κύριο Φαν ο οποίος ε, είναι και τυχερός, αν ήταν εδώ πέρα σήμερα, θα είχε την προσοχή ολόκληρη της Ευρώπης, γιατί όλοι οι υπόλοιποι ε, επικεφαλής κυβερνήσεων πηγαίνουν στα κοινοβούλια τους. Ο κύριος Φαν Ρόμποϊ δεν το έκανε. Και ο κύριος Μπαρόσο και ο κύριος Γιούνκερ σε αυτή την ομάδα. Πού είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν τη συνθήκη, τους λέω, εξ ονόματος της ομάδας μας τουλάχιστον, το τι θα γίνει στην συνθήκη, στην Ευρώπη, στο μέλλον και αν έχουμε επεμβάσει στην εθνική κυριαρχία του προϋπολογισμού δεν γίνεται χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αυτή η κρίση για να συνεχιστεί η υφέρπουσα αποκοινοβουλευτοκοποίηση της Ευρώπης. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό και ελπίζω κυρίες και κύριοι πως αυτό το οποίο θα προκύψει αύριο θα είναι επιτέλους αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Σε τελική ανάλυση δεν έχει τόσο σημασία το περιεχόμενο. Θα πρέπει απλά να δείξουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πως είναι στο ύψος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίφερ Χόφσταθ, για τους φιλελεύθερους και δημοκράτες. Εισαγωγικά θα ήθελα να αναφέρω αυτό το οποίο ε, ανέφερε και ο κύριος Σούλτς. Εγώ σας ανακοινώνω την Πέμπτη θα προτείνω στη διάσκεψη των Προέδρων να καλέσει τον κύριο Μπαρό, τον κύριο Φωνορόμπα και τον κύριο Γιούνκερ να έρθουν να μιλήσουν για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Διότι τους όρισε το Συμβούλιο για να διατυπώσουν προτάσεις για την Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Πιστεύω ότι έχουμε κάθε συμφέρον να έχουμε το Νοέμβριο εδώ παρουσία τους μία συζήτηση. Δεν θα γίνει όπως την τελευταία φορά όπου τελικά έχουμε μία πρόταση και ερχόμαστε πρώτε τελεσμένο. Έχει αποφασίσει ήδη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν μπορεί να επηρεάσει καθόλου τις προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα το ανακοινώνω λοιπόν. Ελπίζω να μα στηρίξουν περισσότερε πολιτικέ ομάδε αν όχι όλε για να γίνει αυτή η συζήτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, αυριανή Σύνοδο μετά από 20 μήνες αντιφάσεων, δισταγμών και ημίμετρων έχω την εντύπωση, την εντύπωση ότι αυτή τη φορά πλέον κατάλαβαν ότι πρέπει να λάβουν μέτρα, μέτρα σε βάθος, ότι χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Ένα συνολικό σχέδιο ώστε πραγματικά να επανέλθει η σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Χρειάζεται επίση ένα ε, χάρτη πορεία, ένα οδικό χάρτη για να υλοποιηθεί αυτό ο στόχο. Ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο του σχεδίου αυτού, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ απλό το περιεχόμενο εδώ στο Κοινοβούλιο και με το Κοινοβούλιο έχουμε μια συντριπτική πλειοψηφία υπέρ ενό ψηφίσματο, ε, το οποίο ψήφισαν πριν από 8 ή 10 μέρε. Ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρει τα μεγάλα ε, μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματο για να έχουμε ξανά σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τίποτε, ούτε να συζητήσουμε κάτι. Έχουμε ιδέε περιλαμβάνοντα ένα σαφέ, ξεκάθαρο ψήφισμα για σε 7 μεγάλε μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Ευρωζώνη. Και νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον εδώ σε αυτή τη συζήτηση και ίσως εσείς κύριε Πρόεδρε όταν φαντάζομαι ότι θα πάτε την Τετάρτη θα είστε εκεί για να κάνετε την παραδοσιακή θα έλεγα εισαγωγή, έναρξη ε, αυτού του ε, Συμβουλίου. Θα σας παρακαλέσω να επαναλάβετε τα επτά σημεία τα οποία ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Δηλαδή βιώσιμη λύση για την Ελλάδα. Είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών γιατί δεν πρόκειται αυτό να επιτευχθεί με εθνικά μέτρα, αλλά χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Επίσης, ε, ενίσχυση του Ταμείου Διάσωσης και τα υπόλοιπα σημεία τα οποία έχουμε συμπεριλάβει στο ψήφισμά μας. Επομένως, και ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, ένα σημείο είναι σημαντικό σε όλα αυτά για τις προσεχείς ημέρες και εβδομάδες. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα, για την οικονομική διακυβέρνηση, μπορούμε να μιλήσουμε για την οικονομική κυβέρνηση, για την οικονομική και φορολογική ένωση που χρειαζόμαστε, για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Όλα αυτά είναι άκρο σημαντικά. Πρέπει να το επαναλάβετε την Τετάρτη στου αρχήγου κρατών και κυβέρνησεων, αλλά είναι γνωστό το βασικό. Το βασικό είναι πώ θα ενισχύσουμε το Ταμείο διάσωση. Αυτό είναι το θέμα για την Τετάρτη, τίποτε άλλο. Για τα υπόλοιπα θα πούν, ορίστε, ναι, ε, θα κάνουμε κάποια πρόοδο ε, για την ε, Σύνοδο Κορυφή του Δεκεμβρίου. Αλλά το θέμα του ουσιώδες είναι αυτό. Πώς θα ενισχύσουμε. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ μίλησε για μπαζούκα. Θα είναι το μπαζούκα πάνω στο τραπέζι. Όταν μιλάμε για τις χρηματοπιστωτικέ αγορές, δεν έχουν απλά κάποια ελαφρά πυρομαχικά. Μιλάμε για βαρέα όπλα. Και μπορώ να σας πω ότι η πρόταση η οποία θα εγκριθεί την Τετάρτη ήδη υπάρχει και κυκλοφορεί στους διαδρόμους. Ενίσχυση του Ταμείου Διάσωσης. Όχι στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στους δρόμους, του Reichstag, της Γερμανικής Βουλής. Ε, Εκεί κυκλοφορεί αυτό το κείμενο το οποίο θα εγκριθεί την Τετάρτη. Και λέγεται σχέδιο όρων και προποθέσεων για τη μεγιστοποίηση τη ικανότητα δανεισμού του EFSF. 3,5 σελίδε που έχουν μέσα του όλε τι λεπτομέρειε για το πώ θα γίνει αυτό. Δεν το έχουμε εμεί στα χέρια μα αυτό. Σε εθνικό επίπεδο κυκλοφορεί αυτό το έγγραφο. Εκεί συζητείται. Όχι στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα. Πρέπει να το διαβάσει κανείς τρεις-τέσσερις φορές και μετά αν καταλάβει κάτι. Και έχω και κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορεί, κύριε Πρόεδρε, να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, διότι πρόκειται για ένα σύστημα με το οποίο θα δώσουμε μια διασφάλιση της άξιος του 20%, ε, γράφεται ήδη στον τύπο, σε όλα τα ομόλογα τα οποία εκδίδονται από χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία, Ισπανία, Ιταλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. 20% θα λάβουν αν δεν μπορεί να ενισχυθεί το Ταμείο Διάσωση, αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη για να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν δεν γίνεται άμεσα στην πράξη να λειτουργήσει μια ενιαία αγορά ομολόγων, τι γίνεται, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά, λέμε τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεχίσουν να εκδίδουν ομολόγα και εμείς οι Ευρωπαίοι θα τους δώσουμε μια εγγύηση της τάξης του 20%. Εγώ αμφιβάλλω για τα πόσο θα λειτουργήσει αυτό. Λοιπόν, 20%. θα μειωθεί το ευρωελληνικό χρέο κατά 60%, θα κουρευτεί κατά 60% και περιμένουμε ταυτόχρονα εγγύηση 20% και όλα αυτά θα καθησυχάσουν τις αγορές τελικά. Α, μακάρι. Μακάρι να λειτουργήσει αυτό. Αλλά αμφιβάλλω. Πολύ αμφιβάλλω. Γιατί νομίζω ότι η μόνη η καλή, η σωστή λύση είναι να δημιουργηθεί μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων στην Ευρωζώνη και για να σωθεί το ευρώ. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος ε, Σαχράντιλ έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου να συνοψίσω τη σημερινή κατάσταση αναφέροντας ε, το γεγονός ότι βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε πίσω. Έχουμε πάει στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, όχι του 21ου. Δηλαδή σε μια Ευρώπη μετά από το 1815, μετά από το συνέδριο της Βιέννης, όπου τότε μιλούσαμε για συνεργασία των δυνάμεων. Γιατί ό,τι και αν λέμε για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, για την κοινοτική μέθοδο, για την ε, ανέβρεση υπερεθνικών λύσεων, τις τελευταίες 15 μέρες δύο άτομα βλέπω που διευθύνουν το θέαμα και που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε μια καγκελάριο και έναν πρόεδρο που μάλιστα τα έψαλε σε έναν πρωθυπουργό και του σύστησε να σιωπήσει. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν και πολύ ευρωπαϊκή. Η κρίση τώρα πάντα το ίδιο συμβαίνει, ότι δηλαδή οι φορολογούμενοι είναι αυτοί που πληρώνουν την ανεύθυνη συμπεριφορά των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παίζουν λες και πρόκειται για καζίνο. Ο φορολογούμενος θα πληρώσει για την ανεύθυνη συμπεριφορά των χωρών που δαπανούσαν δημόσιο χρήμα το οποίο δεν είχαν και τώρα μας προτείνεται να εξευρωπαϊστεί το χρέος, να το αγοράσουμε γιατί λέει διακυβεύεται η σωτηρία της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω πως ε, κανένας δεν διαβάζει τα σχόλια των οικονομολόγων ε, στις εφημερίδες γιατί αύριο καμιά απόφαση δεν πρόκειται να ληφθεί. Απλώς ε, θα κερδίσουμε λίγο χρόνο, θα βρούμε ίσως μια λύση για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια αλλά θα ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό το οποίο δεχόμαστε ε, ανάμεσά μας στους διαδρόμους, αλλά που δεν το δέχεται κανείς δημοσία, ότι το ευρώ δεν είναι για όλους. Ορισμένες χώρες μέλη δεν θα μπορούν να συμμετέχουν γιατί θα πρέπει να υποστούν την υποτίμηση. Όλοι το γνωρίζετε, το συζητάμε στους διαδρόμους, αλλά φοβάστε να το πείτε μεγαλόφωνα. Λοιπόν, λοιπόν και πάλι θα παίξουμε κόντρα στο ρολόι. Ε, είναι μια παραδοσιακή μέθοδος ε, άνετη που όμως είναι πολύ δαπανηρή και λιγότερο αξιόπιστη για τις αγορές. Δεν είναι λύση ενός πολιτικού ανδρός. Ε, ένας πολιτικός άνδρας αντίθετα από έναν πολιτικάντη παρουσιάζει ε, ε, θαραλέες λύσεις ε, και αύριο πραγματικά θα δούμε αν υπάρχουν πολιτικοί άνδρες στην Ευρώπη αν πρόκειται απλώς για αντίδες. Σας ευχαριστώ. Η Ρεμπέκα Χάρμς. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για εμένα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε προκύπτουν δύο πράγματα. Μπορούσε κανείς να δει στο Συμβούλιο με βάση την έκθεση της Τρόικας πως όλα όσα είχαν ληφθεί ως αποφάσεις για την Ελλάδα ήταν λάθος, ό,τι μπορούσε να γίνει λάθος είχε γίνει. Ήδη τον Ιούλιο το Συμβούλιο είχε κάνει ένα κούρεμα της Ελλάδας το οποίο ήδη τότε είχαμε πει πως ήταν πάρα πολύ μικρό. Η επιμονή στην Ελλάδα μονομερός να έχουμε μόνο λιτότητα κατέληξε στην καταστροφή που είχε προβλεφθεί την Ελλάδα δε την σέρναμε από σύνοδο κορυφή σε σύνοδο κορυφή και επιδεινώθηκε έτσι η κρίση, η κρίση του ευρώ και η ευρωπαϊκή άρα κρίση. Και νομίζω πως αυτό το οποίο προκύπτει από την αναβολή του Συμβουλίου είναι πως δεν μπορούμε την Ευρώπη να την καθοδηγούμε μέσω αυτών των συνόδων. Χρειαζόμαστε έναν φόρο σταθεροποίησης και οικονομίες. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων μετά από την τριήμερη διαβούλευσή τους. Εμείς λοιπόν από την επανάληψη της Συνόδου απαιτούμε άλλα αποτελέσματα και να σταματήσει αυτό το συνεχές μοτίβο των συνόδων που είναι πάρα πολύ, λαμβάνουν αποφάσεις πάρα πολύ αργά και πολύ περιορισμένες. Ελπίζουμε το ψαλίδισμα του ελληνικού χρέους να είναι πάνω από το 50% και δεν είναι δυνατόν οι κερδοσκόποι οι οποίοι παίζουν συνεχώς στην χρεοκοπία της Ελλάδας με κρατική εγγύηση να τους κάνουμε πάλι πλούσιους. Αλλά πρέπει να στείλουμε ένα άλλο μήνυμα στην Ελλάδα. Η οικονομία της Ελλάδας, η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των δικών μας μέτρων. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο νοικοδόμησης της ελληνικής οικονομίας και το βάρος πρέπει να δοθεί, λέμε εμείς οι πράσινοι, στην αηφορία. Ξέρω πως δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα αξιόπιστο σχέδιο γι' αυτό. Η απόφαση τώρα για το EFSF, ε, αυτό το μπαζούκα τώρα, ε, αυτός ο όρος ο παρανοϊκός, εμένα δεν μου λέει τίποτα, αλλά πρέπει να πολλαπλασιαστούν τα μέσα του ταμείου αυτού, αλλά όποιος μιλάει και για σταθερότητα θα πρέπει να φροντίσει μέσω των μέσων αυτών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι προϋπολογισμοί. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, από όσο ξέρουμε, πάλι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ αργά η εθνικοποίηση της ευθύνης γι' αυτό θα οδηγήσει εγγυημένα στο ότι η περίπτωση τέξια δεν θα είναι μεμονωμένη αλλά θα επαναληφθεί. Και τέλος είδαμε πώς δεν θα βγει η Ευρώπη από την κρίση. Ναι, να συζητήσουμε για την αλλαγή της συνθήκης, να συγκληθεί μια συνέλευση που θα επιτρέψει και στους Ευρωπαίους να καταλάβουν ποιες θα είναι οι αλλαγές. Αλλά δεδομένης της διάλυσης και των διαφορετικών δρόμων που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και της άμεσης ανάγκης για δράση θα πρέπει να έχουμε θάρρος. Ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία και το προϋπολογισμό θα πρέπει τώρα να αποκτήσει την δυνατότητα να έχει προϋπολογισμούς με αλληλεγγύη και για την οικονομική ανάπτυξη. Και αν δεν έχει το θάρρος για κάτι τέτοιο, δεν έχει την δυνατότητα να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση. Και να σας πω και κάτι από την Γερμανία. Όποιος φοβάται τους ψηφοφόρους του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή κρίση. Τώρα, όταν η Άγγελα Μέρκελ θέλει να... Όταν τη θυμίζουμε τον Χέλμουτ Κόλ και τον Χέλμουτ Σμιτ ε, ή όταν θυμίζουμε στον Κουίντο Βέστερβέλε τον Χέλμουτ Σμιτ, πρέπει πραγματικά να εμπνευστούν και να μπορέσουν και να πούν κάτι στους ψηφοφόρους τους με θάρρος και ίσως τότε να κερδίσουν και τις εκλογές. Αλλά έτσι θα χάσουν και τις εκλογές και πιθανώς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Έχετε μία μπλε κάρτα. Κυρία Χάρμς, ερώτηση προς εσάς. Την δέχεστε? Κυρία Χάρμς, δέχεστε την ερώτηση με την μπλε κάρτα. Μάλιστα. Ο κύριος Χουτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομιλήτρια, αν κατάλαβα καλά, κάποια στιγμή αναφερθήκατε στο θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους και πράγματι είναι ένα από τα θέματα κυκλοφορούν τα σενάρια για 50-60% δεν κατάλαβα ποια είναι η δική σας γνώμη. Θα ήθελα κυρία συνάδελφο επειδή αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις να σας πω ότι το ελληνικό χρέος είναι 360 δις και το κούρεμα κατά 50% δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί κατά 180 δις αλλά θα μειωθεί κατά 25 δις που σημαίνει ότι τη μεγαλύτερη ζημιά θα την υποστούν ελληνικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που θα πουληθούν με χαμηλότερη τιμή. αν αυτά τα στοιχεία είναι αληθή αυτά που λέγω και όχι μαγική εικόνα πείτε μου σας παρακαλώ είναι η γνώμη σας, εξακολουθεί να είναι η γνώμη σας για αυτό το κούρεμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαι πεπισμένη πως εάν δει κανείς την έκθεση της ε, Τρόικας πως πρέπει να γίνει αυτό γνωρίζω πως πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά πιστεύω πως αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν θα τη λάβει κανείς μόνος του. Το σχέδιο του πώς θα ανοικοδομηθεί η Ελλάδα με ευρωπαϊκή βοήθεια, αυτό το σχέδιο πρέπει επίσης να αποφασιστεί και το εύχομαι ως ευρωπαϊκό μήνυμα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες που γνωρίζουν πως θέλουν να, και πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα, ένα τέτοιο μήνυμα αλληλεγγύης δεν έχει δοθεί από καμία από τις συνόδους μέχρι στιγμής στους Έλληνες. Κύριος Λόταρ Μπίσκι της Ενωμένης Αριστεράς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαχείριση της ε, κρίσης γίνεται όλο και πιο χαοτική και αδιάφανη. Το Συμβούλιο έχει μία προ-σύνοδο και μία κύρια σύνοδο. Το ΔΕ Κοινοβούλιο ασχολείται δύο φορές με τα αποτελέσματα της συζήτησης στο Συμβούλιο. Ήδη προδιαγράφεται πως το μεγάλο βήμα δεν θα γίνει ούτε αυτή τη φορά. Οπότε παραμένει μόνο το σχόλιο και Κομισιόν και Συμβούλιο πορεύονται με βάρκα την ελπίδα. Ελπίδα πως τα μέτρα αυτά θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, ελπίδα πως αυτή τη φορά θα ικανοποιηθούν οι αγορές. Αλλά γιατί όσοι στοιχηματίζουν στη χρεοκοπία των κρατών πρέπει να ικανοποιηθούν. Γιατί δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την Ισπανία και την Ιταλία από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται. Μόνο ριζικά μέτρα μπορούν να εμποδίσουν την δυσμενή εξέλιξη για τις χώρες αυτές. Γιατί αλλιώς θα συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και θα συνεχίσει να προτείνει ομπρέλες προστασίας το Συμβούλιο με τα λεφτά των φορολογουμένων. Με οικονομικά τρίκ υποτίθεται πως θα υπάρξει και μόχλευση του EFSF ε, του ποσού των 78 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένας Γερμανός οικονομολόγος μιλάει εδώ πέρα για όπλο μαζικής καταστροφής. Μιλάμε μάλιστα για ένα ποσό 4 3 εκατομμυρίων ευρώ και από ό,τι φαίνεται το κούρεμα του ελληνικού χρέους είναι απόφυκτο και το μόνο ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει το κόστος. Πράγματι θα πρέπει οι διεθνεί τράπεζε να επομιστούν ένα ποσοστό μέχρι 60% αλλά θα πρέπει να εμποδίσουμε τι χρεοκοπίε, Αυτό αφορά ειδικά τι ελληνικέ τράπεζε που απειλείται η ύπαρξή του. Θα πρέπει οι Έλληνε πολίτε μετά από όλε τι κοινωνικέ περικοπέ να ανησυχούν και για τι καταθέσει του και τι οικονομίε του στι τράπεζε. Αντί για μια ομπρέλα προστασίας για τις τράπεζες, χρειαζόμαστε μια ομπρέλα προστασίας για συντάξεις, μισθούς και τις αποταμιεύσεις των πολιτών. Χρειαζόμαστε μια δημόσια τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα δώσει τα απαραίτητα κονδύλια με ευνοϊκά επιτόκια στα κράτη-μέλη και θα αφήσει εκτός τις ιδιωτικές τράπεζες. Χρειαζόμαστε επίσης ένα πρόγραμμα επενδύσεων. Σας ευχαριστώ ο Σύμπροεδρος ε, της Ελευθερίας και Δημοκρατίας, Φραντσέσκος Περόνι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση για την οποία ελπίζω θα βρεθεί μια θετική λύση δείχνει το πόσο ακατάλληλο ήταν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μετά την εισαγωγή του ευρώ. Όλο και μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ των πολιτών, ψηφοφόρων και των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωκοινοβουλίου. Το κοινοβούλιο που θα έπρεπε να εκπροσωπεί τους πολίτες όλο και περισσότερο ε, λαμβάνει αποφάσεις που το απομακρύνουν, που είναι κατά της ε, λαϊκής βούλησης. Υπάρχει το εξής ουσιώδες. Ούτε μπορούμε ούτε πρέπει να υποφεληθούμε από την κρίση για να στερήσουμε τα κράτη-μέλη από την κυριαρχία τους ε, και για να μεταφέρουμε δικαιώματα των πολιτών στην Ένωση. Η Αγγέλικα Βέρτμαν τώρα είναι η επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση εξακολουθεί να υφίσταται και δεν υπάρχει καμία λύση. Η Μίνχενερ, μια εταιρεία αντασφαλίσεων, είπε πως από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει χρεοκοπία της Ελλάδος. Από την άλλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει αποφασιστική πολιτική ηγεσία. Τι συζητάει το Συμβούλιο ακόμα, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα όταν αυτός αρχίζει να δρά από μόνος του από ό,τι φαίνεται η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης τρέχει πίσω από την πραγματικότητα. Μετά από τα όσα μας ανέφερε η Τρόικα την προηγούμενη εβδομάδα, τίθε το ερώτημα το εάν θα αρκέσει το περίφημο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Οπότε από εδώ προκύπτει η έκκλησή μου προς όλους τους υπεύθυνους. Δράστε άμεσα με αποφασιστικότητα και με ενότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εδώ πέρα τελειώνει η συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της